So, dear ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε και καλώς όρισαν οι συνάδελφοι που είναι στην ώρα τους. Οπότε έχετε το σχέδιο μέσα διάταξης. Γιατί το πρώτο σημείο αυτής είναι η έγκριση. Έχετε κάποιο αίτημα για αλλαγή, όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε εγκρίνεται. Σημείο παρθαμών 2 είναι η έγκριση των πρακτικών του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Όσοι συνήθως δεν υπάρχει κάποια ένσταση θεωρούνται τα πρακτικά εγκεκριμένα. Αυτό μέχρι το τέλος της συνδυάσεως. Υπαριθμόν 3. Έχουμε τώρα τις αποφάσεις των συντονιστών. Έχετε λάβει τα σχετικά έγγραφα και για εδώ ισχύει το ίδιο. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, τότε οι αποφάσεις των συντονιστών θεωρείται ότι εγκρίνονται. Τέσσερα. Ως συνήθως μεταδίδουμε στο ίντερνετ τη συνεδρίασή μας ε, και έχουμε πολλούς ενδιαφερόμενους εκτός ε, κοινοβουλίου. Σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή, από το Ταλίν μέχρι τη Ρώμη, από την ε, Λισαβόνα μέχρι το βράδυ. οπότε για αυτό το λόγο να μιλάτε αργά και καθαρά, ούτως ώστε να σας ε, καταλαβαίνουν καλύτερα οι διερμοί και να το έργο τους. Και επίση αυτοί που μας ακούν ε, εκτός ε, κοινοβουλίου και αυτοί να μπορούν να καταλάβουν καλύτερα Έχουμε κάποιο καινούριο συνάδελφο εδώ μέρο Επιτροπή, θα βρίσκεται εδώ, τα πούμε αργότερα όταν έρθει. Οπότε το πρώτο μα θέμα για σήμερα είναι η συζήτηση που αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Και νομίζω όλοι θα έχετε υπόψη το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει μια φιλόδεξη έκθεση για τις σχέσεις αυτές. Η άφατη έχει την πολιτική πτυχή αυτών των σχέσεων και η Επιτροπή του Εμπορίου, η ΙΝΤΑ, ασχολείται με την εμπορική πτυχή των σχέσεων μας με την Κίνα και με μεγάλη μου χαρά σήμερα έχουμε τον πρέσβη της ε, Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Τσάνγκ Μίνγκ. Τον βλέπω εκεί κάθεται, κάτω. Καλώ ορίσατε και έχουμε επίση και τον ε, εισηγητή τη σχετική εκθέσεω, τον κύριο Βίγκλερ, που επίση βρίσκεται στην αίθουσα και συμφωνήσαμε με την ΑΦΕΤ ότι θα επικαλεστούμε το άρθρο 54 του κανονισμού ούτως ώστε όπως ορίζει να αποφασίσουμε όσον αφορά τα του εμπορίου και για αυτά θα έχει λόγο πάνω σε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα Βρίσκονται τώρα στην ε, φάση ε, των διαπραγματεύσεων για εμπορικά θέματα. Βεβαίω η Κίνα είναι ένα ε, μεγάλο και σημαντικό μα εμπορικό εταίρο και όσον αφορά την παγκόσμια συγκυρία και το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου από τη βάση των κανόνων του ΠΟΕ, τα πράγματα είναι πιο σημαντικά από ό,τι στο παρελθόν. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε για το πώς αυτές οι μορικές σχέσεις θα σταθεροποιηθούν. Παρακολουθούμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένα τα της επενδυτικής συμφωνίας. Έχουν γίνει 17 κύκλοι διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα. Άρα βλέπετε ότι Πρόκειται για μακρές και εντατικές διαπραγματεύσεις βεβαίως. Ακούσαμε την ομιλία του Σαντσί στο Νταβός στη συνέχεια του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και σε σχέση με την απόφαση να αλλάξουν οι κανόνες για τις επενδύσεις για τους σχετικούς κανόνες, τους σχετικούς τομείς μάλλον και έτσι τώρα να υπάρχουν νέες δυνατότητες ώστε οι εταιρείε να μπορούν εκεί να έχουν μια παρουσία χωρίς να δεσμεύονται από αυτόν τον κανόνα του 59% ή 49%. Τέλος πάντων θα πρέπει να δούμε κατά πόσο να υπάρχει καλύτερη κατανόηση και περισσότερη αμοιβαιότητα σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις. Και, όπως είπαμε προηγουμένως, όσον αφορά την παγκόσμια συγκυρία, είναι σημαντικό να μπορούμε να συζητήσουμε τις επόμενες φάσεις και να διατηρηθεί ο πολυμερής χαρακτήρας των σχέσεων. Σε δύο εβδομάδες θα πάμε στην Κίνα. Οπότε θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές επαφές με τις αρχές της χώρας και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νομίζω κύριε Πρεσβή είναι η πρώτη σας επίσκεψη εδώ στην Επιτροπή μας. Ίσως και είναι η πρώτη φορά συμμετέχει σε μια ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση εδώ στο Κοινοβούλιο από τότε που μετατεθήκατε εδώ με αυτή την θέση. Οπότε με ιδιαίτερη χαρά μας σας υποδεχόμαστε και τώρα θα σας δώσουμε το λόγο για 10 λεπτά για να μας πείτε τις απόψεις πώς βλέπουν τα πράγματα τόσο αφορά τις σχέσεις μας τις εμπορικές με τη χώρα. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Στρασβούργο και παρακολούθησα εκεί τις ε, εργασίες σας ε, στα άλλα σας κεντρικά ε, κτίρια και σήμερα ήρθα για να βρεθώ μαζί σας εδώ στη κτίρια σας των Βρυξελών για να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις ε, προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή ΙΝΤΑ για την πρόθεση της ε, οικονομικής ε, και εμπορικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Πριν έρθω εδώ, διάβασα το σχέδιο γνωμοδότησης που έχετε εκπονήσει που έχει εκπονήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Είμαι εδώ και στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στην γνωμοδότηση. Πριν μπούμε όμως στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές ιδέες ως βάση για τις συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να τονίσω ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας είναι αμοιβαία επωφελείς από τη φύση τους. Τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Το 1978 όταν η Κίνα μόλις είχε ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα προς τον εξωτερικό κόσμο, το εμπορίο αγαθών μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναρχόταν σε μόλις 4 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών και επενδύσεων ήταν σχεδόν μηδενικό. Μετά από 40 χρόνια, το εμπόριο αγαθών μας ε, ανέρχεται σε πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα το εμπόριο υπηρεσιών έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και οι επενδύσεις σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Μαζί το εμπόριο και οι επενδύσεις μας έχουν αυξηθεί κατά περίπου 250 φορές την τελευταία 40 και Τέτοια ανάπτυξη θα ήταν αδύνατον να γίνει εάν δεν είχε υπάρξει αμοιβαία υποφελή. Τα ωφέλη από το εμπόριο και τις επενδύσεις ε, είναι μεγάλα για την Κίνα αλλά είναι μεγάλα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία της Eurostat ε, δείχνουν ότι το 2017 η αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα έφτασε το 21% της συνολικής αύξησης των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Οι εξαγωγές προς την Κίνα όθησαν ε, τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αύξηση 1,6% περισσότερο από ό,τι πραγματοποίησαν άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να ομολογήσω ότι πράγματι υπάρχουν κάποια ζητήματα στις οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις. Ωστόσο, δεν είναι παρά ένα πολύ μικρό κομμάτι της συνολικής μας συνεργασίας, της οποίας η αξία ανέρχεται σχεδόν σε χίλια δισεκατομμύρια δολάρια. Με ανοιχτά και ομαλά κανάλια επικοινωνία, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιδιώξουν λύσεις μέσω της φιλικής διαβούλευσης. Επίσης πιστεύουμε ότι για να επιληθούν τα προβλήματα πρέπει να κοιτάμε στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Εάν κάποιος αποσυρθεί μέσα σε έναν πύργο προστατευτισμού, σίγουρα δεν θα δει, δεν θα μπορέσει να δει πόσο όμορφη είναι η Άνοιξη έξω από αυτόν. Στραμμένοι λοιπόν προς το μέλλον, δεν είναι δύσκολο να δει κανείς ότι ε, περαιτέρω άνοιγμα της Κίνας θα παρέχει τεράστιες ευκαιρίες για την οικονομική και πολιτική συνεργασία και, και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος μου, ο κύριο Σιτζιμπίνγκ, είπε ότι το άνοιγμα της Κίνας ήταν το κλειδί για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη τα τελευταία 40 χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, είπε ο πρόεδρος, η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας της Κίνας θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο με μεγαλύτερο ακόμη άνοιγμα. Λίγο μετά από το 19ο συνέδριο του κόμματος, η Κίνα εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Στις αρχές του μήνα αυτού, ο Πρόεδρος Σι ανακοίνωσε περαιτέρω μέτρα για σημαντική διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά, για τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για επέκταση των εισαγωγών. Καθώς ε, εμείς υλοποιούμε σταδιακά τα μέτρα αυτά, η Κίνα θα εισέλθει σε μια νέα φάση ανοίγματο προς τον κόσμο. Ο κινέζικος λαός ε, εκτιμά την αξιοπιστία και όταν το λέμε αυτό το εννοούμε έχουμε καθορίσει σαφή διαγράμματα για την αναθεώρηση της αρνητικής λίστας ε, ξένων επενδύσεων. Έχουμε χαλαρώσει τους περιορισμούς ε, για την εγκατάσταση ξένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και έχουμε άρει περιορισμούς ε, για ξένα μετοχικά κεφάλαια σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Ήδη λοιπόν έχουμε αναλάβει δράση. Ένας πρώην αρχηγός ε, κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου είπε η κατεύθυνση είναι πιο σημαντική από τη ταχύτητα. Ένας άλλο φυσικά συνάδελφος δεν συμφωνεί. Λέει ότι η ταχύτητα και η κατεύθυνση είναι εξίσου σημαντικές. Δεν θέλω να τσακωθώ και να αποφασίσουμε αν το κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Αλλά Πιστεύω ότι αυτό ο συνάδελφο θα καθησυχαστεί, αρκεί να δει πόσο αποφασιστικά και με πόσο μεγάλη ταχύτητα κινείται η Κίνα ε, καθώς ανοίγει προς τον υπόλοιπο κόσμο. Οι επενδυτέ ε, συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαίων εμπιστεύονται πλέον το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας, όπως αποδεικνύουν οι επιχειρηματικές τους αποφάσεις. Το 2017 η Κίνα υποδέχτηκε 136,3 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής σε ξένες επενδύσεις. Ποσό ρεκόρ για την Κίνα που την κατέταξε στη δεύτερη θέση παγκοσμίω. Οι άμεσε ξένε επενδύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017, παρότι είχαν μειωθεί ελαφρά σε σχέση με το 2016, εν μέρη λόγω του σχετικά υψηλού αριθμού βάση στα τέλη του 2016, αυξήθηκαν σημαντικά, 24% σε σχέση με το 2015. Μια έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα δείχνει ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα υπήρξαν κερδοφόρες και ότι πάνω από τις μισές από τις επιχειρήσεις αυτές είναι αισιόδοξε για τις μελλοντικές τους πρόπτικες στην Κίνα. Αυτό αποτελεί αδιάσυστη απόδειξη ότι η Κίνα είναι μια ανοιχτή χώρα και ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές το αναγνωρίζουν. Στις οικονομικές και εμπορικές ε, σχέσεις Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι προβλήματα. Για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες ε, απαιτείται ένα σταθερό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα ένα πολυμερές ε, σύστημα εμπορίου βασισμένο σε κανόνες. Έχει ύψιστη σημασία κάτι τέτοιο δεδομένη της ε, αυξανόμενης τάσης του προστατευτισμού και της μονόπλευρης αντιμετώπισης ε, και καθώς εντείνονται οι αβεβαιότητες διεθνώς, μια σταθερή σχέση μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψιστης αξίας. Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικά μέλη του ΠΟΕ αποτελούν ε, στρατηγικούς εταίρους μεταξύ τους. Θα χρειαστεί λοιπόν ε, να σταθούμε ένας δίπλα στον άλλον με μια σαφή στάση και προσέγγιση κατά της μονόπλευρης αντιμετώπισης και του προστατευτισμού. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε το πολυμερές ε, σύστημα εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες και να ακολουθήσουμε ε, μια, αυτή την υγιή ορμή της ε, παγκόσμια οικονομίας. Αυτό είναι κοινή μα ευθύνη. Θα χρειαστεί να δράσουμε μαζί για να κάνουμε κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Ορισμένοι Ευρωπαίοι φίλοι λένε ότι το σημερινό σύστημα λειτουργεί αλλά ότι δεν είναι αρκετά δίκαιο. Η Κίνα είναι πάντα διατεθειμένη να ακούσει τι ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιαδήποτε βελτίωση του συστήματο. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο η μονόπλευρη αντιμετώπιση, ο προστατευτισμός ε, θέτουν σε κίνδυνο τη δική μας ε, ε, πολιτική συνεννόηση προς όφελος βραχυπρόθεσμων συμφερόντων και τα οποία αποδυναμώνουν την οικονομική παγκοσμιοποίηση, υπονομεύουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και πλήττουν τα θεμελιώδη συμφέροντα όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, ε, φέτος ε, ε, γιορτάζουμε τη 15η επέτειο της ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 20η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα τον Ιούλιο. Η Κίνα ελπίζει να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η συνεργασία αυτή, ειδικότερα στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου, να φτάσει σε ένα νέο επίπεδο. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Ίντα θα συνεχίζει να διαδραματίζει έναν θετικό και επικοδομητικό ρόλο. Κύριε Πρόεδρε, εσείς θα επισκεφτείτε την Κίνα τον επόμενο μήνα με τους συναδέλφους σας. Και συγχωρέστε με που δεν θα μπορέσω να έρθω μαζί σας στο Πεκίνο. Σας εύχομαι όμως ε, ένα καλό ταξίδι και είμαι βέβαιος ότι αυτή η εμπειρία από πρώτο χέρι θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την Κίνα καλύτερα. Ελπίζω ειλικρινά ότι όλο και περισσότεροι συναδελφοί σας θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Κίνα, να μάθουν τη χώρα μου, να τη γνωρίσουν από κοντά. Με την αμοιβαία κατανόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μπορούμε να μεγαλώσουμε την πίτα ώστε η μερίδα που αντιστοιχεί στον καθένα τους πολίτε μας να είναι μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση με όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, παρουσίαση και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συζητητή μας κύριο Βίνκλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ εξοχότατε ε, πρέσβη, κύριε Πρέσβη για τα σχόλιά σας. Ε, πράγματι είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ε, αυτές τις συζητήσεις, διότι και αύριο θα έχουμε μια συζήτηση σχετικά με τις ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και επίσης ε, ε, βλέπουμε ότι ο κύριος πρέσβης τόνισε τις σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Κίνα. Η αποστολή μας θα πάει στη Σανγκάη και στο Πεκίνο σύντομα ε, και εκεί λοιπόν θα συζητήσουμε τις ε, απόψεις των Ευρωπαίων ενδιαφερόμενων ε, μέρων αλλά και θα έχουμε κατατόπους εμπειρίες σχετικά με το τι ακριβώς συνεισφέρει στο διμερές μας εμπόριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Εξοχότατο για την υποστήριξη που παρέχει στην αποστολή, στην της ΙΝΤΑ. Στην, στο σχέδιο γνωμοδότησης βέβαια υπάρχει υπάρχει ελάχιστος χώρος ε, για να κάνω κάποια ε, σχόλια και γι' αυτό τον λόγο ε, η συζήτηση αλλά και οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και οι προτάσεις από τους συναδέλφους μου στην Ίντα θα εμπλουτίσουν το, την γνωμοδότηση της Ίντα προς την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ορισμένα από τα βασικότερα σημεία εντάχει όσον αφορά την ε, γνωμοδότησή μου έχουν ως εξής. Ε, πρώτον, αναφέρομαι ε, στην συμφωνία, στην συμφωνία για τις επενδύσεις. Βρισκόμαστε στον 17ο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος μόλις ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Έχει υπάρξει ε, πρόοδος ε, και υπάρχει πρόοδος, όμως ε, η πρόοδος αυτός, αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να συζητήσουμε στην Επιτροπή τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Εμείς εδώ στην Επιτροπή καλούμε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στην στην αγορά και να υπάρχει πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιριών στην ε, Κίνα ε, και ε, επιθυμούμε να υπάρχει μια αντιμετώπιση μη διακρίσεων προς τις εταιρείες μας και επίσης θέλουμε να υπάρχουν και ρήτρε βιώσιμης ανάπτυξης στην συμφωνία. Επίσης έχουμε την συμφωνία μια ζώνη ένας δρόμος της Κίνας όπου ε, ζητούμε να υπάρχει διαφάνεια σε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Ε, θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και καλούμε να υπάρχει μια πιο ενεργή συμμετοχή της Κίνας σε αυτό το θέμα. Επίσης υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν είναι καινούργια και τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν. Για παράδειγμα, ε, το ε, ζήτημα ε, το οποίο αφορά την... το πλεόνασμα και επίσης τα ζητήματα των γεωγραφικών ενδείξεων. Επίσης, το 2015 ε, ξεκίνησε μια επίση πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά του Προέδρου ε, Ξή στην ε, Κίνα και φυσικά βρισκόμαστε σε άμαυση επαφή με τις εταιρείε μας μέσω του εμπορικού μας επιμελητηρίου στην Κίνα. Επίσης υπάρχει η ανησυχία ότι ε, για την ώρα δεν υπάρχουν ε, σημαντικές ε, λύσεις όσον αφορά τις τεχνολογικές μεταφορές. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία τα οποία θέλω να αναφέρω. Βέβαια θα πρέπει ε, να ε, συζητήσουμε ε, και για τα, τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε στην Κίνα και θα πρέπει να συζητήσουμε και για κάτι άκρως ενοχλητικό όταν λοιπόν ζητάμε από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα σχετικά με τις τάσεις που παρατηρούν στην κινέζικη αγορά τότε δυστυχώς αναφέρουν αρνητικές και όχι θετικές ε, τάσεις ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε με ειλικρίνεια ε, και αμοιβαίο Επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά τα όσα, χαιρετίζω τα όσα είπε ο πρέσβης και ε, όσα αφορούν τις υποσχέσεις ε, και τις διακηρύξεις που έγιναν από τον ε, πρόεδρο της Κίνας πρόσφατα στο φόρουμ του ΜΟΑΟ για την Ασία που έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες έγιναν υποσχέσεις για το άνοιγμα της κινέζικης οικονομίας, ε, κάτι το οποίο επανέλαβε ο πρόεδρος της ε, Κίνας. Ε, ολοκληρώνοντας λοιπόν, χαιρετίζουμε αυτές τις δεσμεύσεις, είναι πολύ σημαντικές δεσμεύσεις, φαίνονται αρκετά υποσχόμενες όμως ε, ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε όλες αυτές τις ε, δεσμεύσεις ε, να αρχίσουν να λειτουργούν και να αποφέρουν αποτελέσματα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν ε, θα ήθελα να πω αν κάποιος ε, με ρωτούσε να πω σε μία πρόταση, την προσωπική μου πρόταση ε, για την ευρωπαϊκή προσέγγιση στις ευρωσυνικές σχέσεις θα έλεγα ότι θα πρέπει πάντοτε να στοχεύουμε στην συνεργασία και πιστεύω ότι οι συναντήσεις μας και οι συζητήσεις μας και αύριο θα συμβάλλουν προς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλα. Και τώρα έχουν ζητήσει το λόγο συνολικά 10 συνάδελφοι και έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Και ε, φυσικά ε, και η Κομισιόν, ο Πρόεδρος αλλά και ο κύριος Βίνκλα θα πρέπει να έχουν ε, το λόγο και γι' αυτό το λόγο σας δίνω στον καθένα 1,5 λεπτό. Η κυρία Μόσκα λοιπόν είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρέσβη για την παρουσία σας και για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για τα τελευταία σας ε, σχόλια στα οποία συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά την ε, κοινή κατανόηση, συνεννόηση και συνεργασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε ιδιαίτερως όσον αφορά το πολυμερές περιβάλλον. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Εσείς υπογραμμίσατε πόσο έχουν αυξηθεί οι συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Παρότι λοιπόν υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας, παραμένουν πολλές προκλήσεις. Οι επενδύσεις πράγματι έχουν αυξηθεί, αλλά από το 2012 έχουν σημειώσει ε, σταθερή σταδιακή μείωση Τρει είναι οι ερωτήσει που θέλω να σας απευθύνω λοιπόν σε σχέση με το αίτημα το δικό μας περί αμοιβαιότητα και level playing field. Από τη μία πλευρά αναφέρατε εσείς ε, τις κινέζικες πρωτοβουλίες όσον αφορά την προστασία των δικαιωματών ε, διανοητικής διεκτησίας και τη ε, μεταφορά τεχνολογιών. Τι ακριβώς κάνετε για να ενεργοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες. Δεύτερον, για τις δημόσιες συμβάσεις, για το public procurement και εδώ χρειάζεται να μας δώσετε κάποιο μήνυμα μέγιστης αμοιβαιότητας για τις δικές μας επενδύσεις και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Τρίτον, χρειαζόμαστε καλύτερη διακυβέρνηση για την πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος» ε, ως ένδειξη ε, μεγαλύτερων δυνατοτήτων αμοιβαιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ECR, κύριε Μέτλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Πρέσβε που ήρθατε για να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα στις σχέσεις μας με την χώρα σας. Ε, αυτά που ακούσαμε είναι θετικά και θέλω να σας πω και Πρέσβε τα εξής δύο. Αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το σχετικό δίκαιο στην Κίνα και τι κάνει η κυβέρνησή σας ε, για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει ούτως ώστε να υπάρχει το δέον επίπεδο προστασίας. Αν θέλετε, πέστε μας τι ισχύει για τα ξένα δικαιοπνευματική της στη χώρα σας. Τι είναι επίση στο μεταπηδικό τομέα όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας. Τι θα γίνει αν ξέρετε λεπτομέρειες να μας πείτε. Και αυτή η πρωτοβουλία που έχει αναπτυχθεί αποτελεί και για τις δύο πλευρές ευκαιρία. Οπότε με το διάλογο να δούμε πώς θα μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε τις ευκαιρίες και να συνεργαστούμε. Άλτε, χείρισου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αξιότιμε πρέσβη. Αρχικά, ε, προς τον κύριο Βίνκλερ θα ήθελα να πω ευχαριστώ ε, πολύ ε, για την ε, γνωμοδότησή σας. Είναι πολύ καλή. Θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες σε διάφορα ζητήματα για να το κάνουμε το κείμενο πιο ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πολύ παρόλα αυτά. Για εμάς τους φιλελεύθερους το διεθνές εμπόριο, οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Πιστεύουμε ότι συνεισφέρουν στην ευημερία και στην συνεργασία Βέβαια υπάρχουν και κάποια πλαίσια, όπως είναι το ζήτημα της αμοιβαιότητας, το οποίο αναφέρθηκε επανειλημμένως ε, σήμερα, ε, και το ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων και του ε, δίκαιου ανταγωνισμού, τα οποία αναφέρθηκαν ήδη στην γνωμοδότησαν, όπως επίσης και τα ζητήματα του πλεονισμού, ειδικά στον τομέα χάλιβα ε, πάνω σε αυτά λοιπόν θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε. Το ε, θέμα όμως που το οποίο με απασχολεί εμένα ιδιαίτερος είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Το το τι θα διασφαλιστεί αλλά και το πώς εφαρμόζεται στην Κίνα αλλά και το ε, ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας και κύριε Πρέσβη ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να μας αποσχολήσει είναι ε, το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή η ε, Κίνα κάνει διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία με, τον, με το Hong Kong. Έχετε κάποιες προφορίες πάνω σε αυτό για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τους πράσινους ο Κλάους Πούχλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γρήγορα για να τελειώσω εν καιρό. Σήμερα η Κίνα είναι ένας ε, πολύ σημαντικός οικονομικός παγκόσμιος ε, παράγοντας ε, είναι μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, παρόλα αυτά όμως ε, μας λείπει το να, να παίξει ένα σημαντικό ε, ρόλο στον τομέα. Λυπούμαστε για τις τελευταίες νομοθετικές αποφάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι η Κίνα δεν είναι ανοιχτή σε άλλες ιδέες, σκέψεις, αλλά και κεφάλαιο. Οι αποφάσεις των μελών του κόμματος να συμμετέχουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι μονάχα μερικά από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Αν δούμε ε, τις ε, σχέσεις με την Κίνα, η αμοιβαιότητα που αναφέρθηκε επανειλημμένως ε, είναι κατά τη γνώμη μας ένα σοβαρό θέμα, διότι η αμοιβαιότητα δεν θα πρέπει να είναι ένα θέμα για τη δημιουργία επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στρατηγικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φιλελεύθερη δημοσιογραφία Δημοκρατία και την υπεράσπιση αυτής η ε, διμερής ε, συμφωνία επενδύσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια ε, ρήτρα βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει όλα αυτά να συμπεριληφθούν και να είναι εφαρμόσιμα, δηλαδή διαφορετικά σε σχέση με τα ως τώρα, ως τις, ως τώρα συμφωνίες, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένα κεφάλαιο για την εφαρμογή αυτών. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την ΓΚΟΕ, ο Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ε, τον εξοχότατο τον ε, πρέσβη της Κίνας που βρίσκεται εδώ μαζί μας για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και εγώ υποστηρίζω και ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Βίνκλερ, για αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο. Πιστεύω ότι δίνει μια καλή κατεύθυνση. Και μπορώ να συμφωνήσω ενίοτε είναι σημαντικότερο να συζητά κανείς και να συμφωνεί το προς τα που κινείται η συνεργασία μας, ε, η εμπορική, η οικονομική αυτή συνεργασία, παρά να συζητά περί ταχύτητας. Διότι όταν οι δύο μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο, ε, όταν μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους και 560 εκατομμύρια ανθρώπους και αυτοί συμφωνούν για την παραγωγή, την κατανάλωση, τις συνθήκες οργάνωσης ε, των όλων συναλλαγών, αυτό επηρεάζει σημαντικά τις καθημερινές ζωές ε, των πολιτών. Μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε για νούμερα και για εκατομμύρια, αλλά αν ένα δισεκατομμύριο πολίτες ε, έχει την εντύπωση ότι δεν τον συμφέρει όλη αυτή η συναλλαγή, τότε τους χάνουμε από το πλευρό μας δεν θα συμμετέχουν στη μελλοντική οργάνωση και δομή. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να συμφωνήσουμε και να συζητήσουμε στον ΠΟΕ. Να έχουμε δηλαδή ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα που δεν θα οδηγεί σε μάχες για βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα, αλλά θα επιλαμβάνεται του μέλλοντος ανθρωπότητας. Και καθώς μιλάω για ανθρωπότητα, θελήσω και εγώ να προσθέσω κάποια, κάποιες παρατηρήσεις ε, στην έκθεση αυτή για μια ελπίζουμε καλύτερη ε, συνεργασία και για περαιτέρω εξέλιξη αυτής της έκθεσης της ΣΥΝΤΑ. Για την EFDD τον λόγο έχει η κυρία Τιτσιάνα Μπέγκιν. Πρόεδρε ευχαριστώ και συνάδελφοι και εγώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη γιατί ήρθε στην συνάντησή μας πρόκειται για ένα εμπορικό εταίρο πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη. Αν θέλουμε όμως να έχουμε υγιείς οικονομικές σχέσεις, βιώσιμες και κερδοφόρες για τις δύο πλευρές, θα πρέπει να δούμε κάποια σημεία. Ε, ωραία, καλό είναι που ήρθε εδώ ο κύριος Παύλης για να τα συζητήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, παραγωγή, τι γίνεται με ε, τα όσα ισχύουν στον τομέα του Χάλιβα. Δεν είναι πάντοτε τα πράγματα τόσο ε, διάφανα με την παροχή των ε, ποδηλάτων και όχι μόνο και οι τελευταίες εβδομάδες επίσης φάνηκε ότι χρειάζεται να δεσμευθεί η Κίνα όσον αφορά την υπερπαραγωγή. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το dumping, τι γίνεται με τα εμπορικά τρίγωνα τα οποία ισχύουν και με άλλες χώρες και να καταπολεμηθούν οι παραποιήσεις και οι και επίσης θα πρέπει για τα προϊόντα διατροφής να δούμε τι θα ρυθμιστεί για τα τυριά από Ιταλία και Γαλλία πολλές φορές ε, για λόγους που δεν είναι σαφείς μπλοκάρονται στα κινέζικα σύνορα αυτά τα εμπορεύματα. Να δούμε τι γίνεται με τις ενδείξεις και εκεί υπάρχει θέμα στο οποίο πρέπει να βρεθεί μια ξεκάθαρη λύση εμείς ως κόμμα νέα θέλαμε να υπάρχει μια προσέγγιση, να προστατεύονται τα προϊόντα μας. Θεωρούμε πάντως ότι είναι ευκαιρία και όχι κίνδυνος η χώρα, αλλά ήρθε βέβαια και η στιγμή τούτο να αποδειχθεί ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και τώρα τα υπόλοιποι συνάδελφοι. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις Νομίζω ότι ακόμα επικρατεί σύγχυση στην Ένωση όσον αφορά την Κίνα και το μέλλον. Μάλλον γιατί δεν μπορέσαμε ακόμα να χωνέψουμε την γεωπολιτική σημασία της ε, Κίνας και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική και η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία που έχει αναλυθεί. Θα πρέπει επίσης να είμαστε ευέλικτοι στις σχέσεις μας. Και για το 16 1 για κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αυτό είναι σημαντικό. Ε, Εμεί το κρατεχόμαστε, αλλά δεν είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά και για κάποιε μεγάλε δυτικέ χώρε. Τώρα, όσον αφορά το εμπόριο, έχουμε 20 κράτη-μέλη που όπως η Γερμανία έχουν ως κύριο εμπορικό εταίρο την Κίνα, βλέπετε επομένως την στροφή που έχει σημειωθεί στα γεωπολιτικά. Άρα, να ξανασκεφτούμε τις σχέσεις μας με την ε, Κίνα. στρατηγικό εταίρο είναι εκεί, Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πούμε σε όλα ναι, αλλά να έχουμε ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, όσον αφορά μια ισόρροπη σχέση, όσον αφορά τι εμπορικέ σχέσει. Και ε, άρα με πνεύμα συνεργασία θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και πάλι ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη που ήρθατε εδώ για να συζητήσουμε. Και τώρα ο κύριο Ντάρτμουθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Α, να το τρώω το άναψε. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη και εσά και το επιτελείο σας που ήρθατε και έχουν εδώ τα εξή σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν τη συζήτηση. Το 2016 το έλλειμμα και με το Βασίλειο είναι 175 δις ευρώ. Και επίσης βλέπω εδώ από το ΕΓΙΣ που είναι πανευρωπαϊκό εργαλείο ας πούμε στην, στην ε, μεταπηγή βιομηχανία ότι εσείς χρησιμοποιείτε πάρα πολλά ε, κρατικά και ε, ενισχύσει και έχετε τον ταμικό στρατηγική ότι καταβλέπετε την αμυντική βιοκρισία και άλλα. Και στην Ευρώπη κάθε μέρα χάνονται θέσει εργασία ω αποτέλεσμα των δικών σα πρακτικών. Και στη συνέχεια αναφέρεται ότι σχεδιάζεται μία εντυπωσιακή άνοδος στην παραγωγή σε 10 τομείς, αναβάθμιση τη βιομηχανίας σας και αυτό επίση θα σημαίνει εθνικοποίηση βασικών τομέων της βιομηχανία. και αυτό βέβαια μαντάτα για τις ξένες επιχειρήσεις. Τέλος αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα, ε, θα κανονίσουν έτσι τις εισαγωγές τους που αυτό θα πλήξει και την Ευρώπη. Τι λέτε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Είμαι. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ με όλους όσοι έλαβαν τον λόγο προηγουμένως για να σταθώ στα εξή δύο σημεία που κανείς δεν ενέφερε. Εν ώψη των μελλοντικών εξελίξεων και για το τι κάνει η χώρα σας όσον αφορά την τεχνητή ευφυΐα, τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα προστατεύσετε τον ιδιωτικό βίο, τα δεδομένα, πώς θα φροντίσετε να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια για αυτά τα στοιχεία τώρα για τον ΠΟΕ. Είναι θέμα προτεραιότητας, είναι θέμα παγκόσμια σημασία. Και όλοι θέλουμε, όχι μόνο να τον σώσουμε τον ΠΟΕ, να τον βελτιώσουμε και θέλουμε να έχει πολυμερή χαρακτήρα. Φυσικά και με αυτά δεν συμφωνεί ο Τραμπ. Και για πέστε μας, εσείς, θα, πώς θα βοηθήσετε να είναι πολυμερής ο ΠΟΕ ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εμπόριο το οποίο διέπεται από κάποιους κανόνες. Τελευταία, πώς βλέπετε το θέμα των μελών που δεν έχουν εκπρόσωπο ή που εκπρόσωπό τους το δευτεροβάθμιο ιδιωτικό όργανο ε, έχει λήξει η θητεία. Ε, Βεβαίω και θέλουμε να διαλέξουμε μια πολιτική συνεργασία και όχι αντιπαράθεση. Και τώρα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε λεπτά. Μάρκο Ρουλό. Thank you. Good afternoon. Um... Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να ε, συγχαρώ ε, τον εισηγητή για την ε, πρόταση που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία των σχέσεων, των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Η ε, Κίνα είναι ένας ε, σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ένωση, ο δεύτερος ε, μεγαλύτερος και παρά τις κάποιες διαφορές, το έλλειπα, την έλλειψη αμοιβαιότητας και τις ίσες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην Κίνα. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να βρούμε την, ε, ε, την ισορροπία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και αναγνωρίζουμε σε αυτό το πλαίσιο ότι πιο ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Έχουμε ακούσει ε, για ε, αρκετά ε, χρόνια και το ακούσαμε και σήμερα από τον εξοχότατο πρέσβη της Κίνας την βούληση να υπάρξουν βαθιές μεταρρυθμίσεις στην αγορά και την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματα όπως μόλις επέ, επιβεβαίωσε ε, ο ε, πρέσβης ε, και να ανοίξει περαιτέρω την οικονομία της και να παίξει έναν σταθεροποιητικό ρόλο στα, στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται το, εμπορ... το διεθνές εμπόριο. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να παραλείψουμε αυτά τα λόγια. Βέβαια πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν. Ε, είναι πολύ ε, σημαντικό η Κίνα να τηρήσει τις υποσχέσεις της όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις όπως είναι για παράδειγμα οι, οι διαπραγματεύσεις για τις επενδυτικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαπραγματεύσεις, ε, ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο ε, Πεκίνο και ακόμα αξιολογούμε ε, την συνολική αξιολόγηση των των κανόνων που πηγαίνει αργά ακόμα ε, δεν είναι αντίστοιχο των προσπαθειών και της δέσμευσης από τη δική μας ε, πλευρά ε, και ελπίζουμε λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να επιταχυνθούν υπάρχει έντονο αίσθημα ότι η Κίνα θα πρέπει να αρχίσει να τηρεί τους ε, κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ε, με βάση το ε, παρελθόν της τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα και θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το πλαίσιο. όπως η Κίνα έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον ΠΟΕ και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσουν κινήσεις οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο προς την εφαρμογή ε, των δεσμεύσεων ΠΟΕ ή αποτελούν παραβίαση ε, των ε, δεσμεύσεων ΠΟΕ. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η υπόσχεση της, ευρωπαϊκή της Κίνας να τηρήσει το εμπορικό πλαίσιο είναι κάτι καλό. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει αυτό είναι αποτρέποντας στρεβλώσεις στην αγορά και αυτό η Κίνα μπορεί να το κάνει αντιμετωπίζοντας προβλήματα όπως είναι το πλεόνασμα το οποίο αναφέρθηκε από πολλά μέλη παρέχοντας επίσης την ίδια πρόσβαση στην αγορά της που έχουν οι κινέζικες ε, ε, εταιρείες ε, αλλού. Ένα παράδειγμα αφορά ε, την ε, ε, τήρηση των προτάσεων, των συστάσεων όσον αφορά το, τα πλεονάσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες. Είναι σημαντικό ότι η υπεράσπιση του, του πολυμερούς εμπορικού πλαισίου είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη κανόνων που θα καλύψουν τα κενά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτό αφορά ζητήματα όπως είναι οι ε, βιομηχανικές επιδοτήσεις, ε, η ε, προστασία επιχειρήσεων. Η συνεργασία με την Κίνα λοιπόν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα άκουσα μέλη ε, τα οποία αναφέρω, αναφέρθηκαν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και αυτά ε, συμπεριλαμβάνονται ε, στην στρατηγική μας για την πρόσβαση της αγοράς ε, και ε, γίνονται διάλογοι σε όλα τα επίπεδα με την Κίνα ε, και βρίσκονται πολύ υψηλά στις προτεραιότητες μας. Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν χαίρεται που, τον, που καλωσορίζει τον Υπουργό Εμπορίου και που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για ζητήματα διμερούς εμπορίου ε, και σε αυτό ε, το πλαίσιο έχουμε ε, και του χρόνου, τον Ιούλιο μάλλον που θα γίνει η επόμενη συνάντηση για τις σχέσεις Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα υπάρχει καλή συνεργασία πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Σας δίνω τώρα ξανά τον λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο κατάλογος που ουσιαστικά δείχνει πόση σημασία δίνεται στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Επιτρέψτε μου να απαντήσω την ερώτησή σας ε, στα κινέζικα. Αυτό θα μας βοηθήσει ε, καλύτερα για να είναι και πιο σαφές η μετάφραση. Ε, ε, η πληροφορική είναι προτεραιότητα για την Κίνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή είχαμε 16 γύρους συνομιλιών και διάφορες διασυνοδικές συναντήσεις. Την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο οι συναδελφοί μας ε, σε επίπεδο εργασίας ε, είχαν μια συνάντηση και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Αλλά απομένουν πολλά να γίνουν. Φυσικά και οι δύο πλευρέ θα συνεχίσουν τι σκληρέ προσπάθειε για τι διαπραγματεύσει ε, και από τι παρατηρήσεις σα ξέρω ότι έχετε κάποιε επικρίσεις όχι μόνο κατά τη κινέζικη ε, κυβέρνηση και η κινέζικη κυβέρνηση, συγγνώμη, και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζουν τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Uh, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κίνα θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επιτεχυνθούν οι συνομιλίες ε, να, μειωθούν, να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο μερών, να προσπαθήσουμε να βρούμε υλοποιήσιμες λύσεις σύντομα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις επί του κειμένου και να γίνει μια ανταλλαγή μιας ενεργού λίστας. Όσον αφορά τις κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη, συμφωνώ με έναν από τους προηγούμενους ομιλητές που είπε ότι η Κίνα αποτελεί ένα χώρο ευκαιρίας ε, για την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, οι κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη δεν είναι τόσο μεγάλες, αντιστοιχούν μόνο στο 2% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Äh, uh, Αλλά οι κινέζικες επενδύσεις εδώ στην Ευρώπη ε, έχουν βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία και έχουν δημιουργήσει τοπικά θέσεις εργασίας example, not Για παράδειγμα, όχι μακριά από τις Βρυξέλλες ε, έχουμε τα εργοστάσια της Volvo, ένα ε, εξαιρετικό παράδειγμα κινέζικων επενδύσεων στην Ευρώπη, που βοήθησαν να βελτιωθούν οι επιδόσεις ε, της επιχείρησης και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Uh, και το τρίτο που ήθελα να τονίσω είναι οι επενδύσεις, ε, οι κινέζικες επενδύσεις ε, στην Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Κίνα. Βασίζονται και αμφότερες οι πλευρές ε, στις των αγορών. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει και δεν το έχει πράξει μάλιστα. Κατά την άποψή μου αυτή η επενδυτική συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και από τις δύο πλευρές. για την πρωτοβουλία «Μια ζώνη, ένα δρόμο, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτέ για την προσοχή τους. Συμφωνώ ότι η πρωτοβουλία μια ζώνη ένας δρόμος ε, θα πρέπει να είναι διαφανής, να συμμορφώνεται με τους παγκόσμιους κανόνες και τις ε, αξίες και τους κανόνες των αγορών και να βοηθά και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και ο λαός της Κίνας και ο πρόεδρος και εγώ ως πρέσβης έχουμε αναλάβει και επαναλάβει τις ίδιες δεσμεύσεις. 呢是中方为国际社会，呃，在呃几年前世界金融危机的背景之下，来为世界经济增添活力而提出的一个建议倡议，呃，来为国际社会提供一个平台。And also I want to emphasize. Θα ήθελα επίση να τονίσω για την πρωτοβουλία αυτή ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα που προσφέρει η Κίνα

Uh, it does not mean that China is offering. Η ε, Κίνα δεν προσφέρει μια πίτα έτοιμη στην Ευρώπη, την οποία μοιραζόμαστε μαζί. Ε, απαιτείται συμμετοχή όλου του πλανήτη και πρέπει να προωθηθεί η συνδεσιμότητα και να ενισχυθεί η παγκόσμια οικονομία. Ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η Ευρώπη είναι φυσικός εταίρος της Κίνας ε, στην πρωτοβούλια ένας δρόμος, μια ζώνη. Πολλοί αναφέρθηκαν στο χάλιβα και στο αλουμίνιο και στο ε, πλεόνασμα παραγωγής. Το πλεόνασμα παραγωγής ε, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δεν αφορά μόνο τον τομέα του αλουμινίου και του χάλιβα. Η πρόκληση αυτή λοιπόν δεν αφορά συγκεκριμένα την Κίνα. Είναι ένα σύνηθες πρόβλημα ε, κατά τη... που προκύπτει από την οικονομική ανάπτυξη. πλεονάσμα παραγωγικότητας είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα οικονομικό. Οφείλεται ουσιαστικά στην παγκόσμια οικονομική ύφεση και στη συρρήκνωση της παγκόσμιας ζήτησης μετά από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Για την Κίνα, η παραγωγή χάλιβά μας. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της ε, καταναλώνεται εγχώρια. Λιγότερο από το 15% του χάλιβά μας εξάγεται. και ουσιαστικά η Κίνα δεν ενθαρρύνει τις εξαγωγές χάλιβα διότι ο τομέας αυτός είναι ενεργοβόρος και τα ενθαρρύναμε τις εξαγωγές θα σημαίνει ότι θα θυσιάζαμε πολλούς σπόρους και το περιβάλλον είναι υπερβολικά υψηλό τίμημα για μας. 几十万的职工的分流安置，这是非常艰巨的一个任务。And και η κινέζικη κυβέρνηση πάντα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και ειλικρίνεια την, το πλεόνασμα παραγωγής του Χάλιβα. Από το 2016 ε, η Κίνα έχει περικόψει 150 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ε, παραγωγής, ε, το οποίο σημαίνει περικοπή πολλών θέσεων εργασίας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή για μας. Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας κατά πέντε λεπτά. Έχετε ε, μιλήσει για το διπλάσιο χρόνο από ό,τι υπήρχε διαθέσιμο. Σας παρακαλώ ε, να επιταχύνετε. Uh, a few words on subsidies.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί οι ευρωβουλευτές ε, έκαναν τόσες πολλές ερωτήσεις. Ε, αν έχει τελειώσει ο χρόνος μου θα χρειαστεί να σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Είμαι πεπισμένο ότι αυτό δεν θα είναι και το τέλος της συζήτησης, απλά μια αφιτηρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και για να κλείσουμε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ε, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για τις ε, προτάσεις. Και πιστεύω λοιπόν ότι τις επόμενες ημέρες θα συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες και η γνωμοδότησή μας θα είναι η καλύτερη δυνατή. Εντάχει δύο θέματα ε, πρώτον, όσον αφορά το, τη συζήτηση με τους συναδέλφους, ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά ειλικρινείς ε, ε, για να συζητάμε ξεκάθαρα σχετικά με προβλήματα και καταστάσεις ε, που ε, δεν ε, αποτελούν το κοινό μας όραμα όπως αφορά το ζήτημα συνεργασίας 16 συν 1. Θα πρέπει να το συζητήσουμε ξεκάθαρα. Είναι μια κατάσταση, δεν είναι τόσο ε, απλό. πρέπει να σεβαστούμε επίσης και στο πλαίσιο της συνεργασίας 16 ε, 1 τους κανόνες που υπάρχουν και να είμαστε διαφανείς. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι κανόνες διότι έτσι θα έχουμε μια συνεργασία που θα είναι κομμάτι της συνεργασίας συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κίνας ε, και φυσικά το λέω αυτό ερχόμενος από μια χώρα που είναι ε, τμήμα αυτής της συνεργασίας 16 1. Και τέλος κύριε Πρέσβη ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις στα ερωτήματα των συναδέλφων. Κλείνοντας θα ήθελα να παραθέσω τις ε, τα όσα έχει πει ε, το εμπορικό μας επιμελητήριο στην ε, Κίνα για την αναφορά του, του 2017-18 ή ένα μεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λοιπόν θεωρούν ότι δεν αντιμετωπίζουν την ίδια βοήθεια όπως οι κινέζικες εταιρείες. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος ε, και ε, θα πρέπει να επιληθεί για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη και ε, καρποφόρα συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Στις 25 Απριλίου το μεσημέρι μέχρι τότε μπορείτε να καταθέσετε τις τροπολογίες. Θα έχουμε μια ψηφοφορία κατά τον Μάιο για να δώσουμε την ε, γνώμη μας προς την ΑΦΕΤ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε ε, Πρέσβη και εδώ τελειώνουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης πριν πάμε στο επόμενο και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καλωσορίσω έφυγε ένα νέο μέλος το οποίο όμως δεν είναι άλλο ανάμεσά μας. Πάμε στο έκτο σημείο της ημερήσιας διάταξης λοιπόν που αφορά την ε, κατάσταση σχετικά με τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στις εισαγωγές ε, χάλιβα και αλουμίου. Βρισκόμαστε σε μια αρκετά σοβαρή κατάσταση όπως γνωρίζετε. Ο πρόεδρος ε, Τραμπ ε, στις 22 Μαρτίου ανακοίνωσε ε, νέους δασμούς 25% στον χάλιβα και 10% στο αλουμίνιο και με βάση την πράξη για την προώθηση του εμπορίου σημείο 232 του 1962, το οποίο επιτρέπει τον πρόεδρο να λάβει μέτρα σε περίπτωση που απειλείται η εθνική ασφάλεια της χώρας. Ακόμα και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, υπήρξαν ανησυχίες για την χρήση αυτής της ε, παλαιάς ε, πράξης. Παρόλα αυτά όμως ο πρόεδρος το έκανε για, τις Ηνωμένες, για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες υπήρξαν εξαιρέσεις παρόλο ε, που δεν ήταν ε, ξεκάθαρο ποιοι ήταν οι όροι ε, για τις εξαιρέσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως η Ιαπωνία για παράδειγμα. Παρόλα αυτά λάβαμε αυτές τις εξαιρέσεις και υπήρξε μια ξεκάθαρη δήλωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε υπό πίεση την μορφή των εμπορικών μας σχέσεων. Αυτή λοιπόν ε, είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση όπως την αντιλαμβάνουμε. Η ε, εξαίρεση αυτή όμως ε, λήγησε μερικές ημέρες την 1η Μαΐου και για να αλλάξει αυτό θα πρέπει ο πρόεδρος να κινηθεί πάνω σε αυτό. Θα το συζητήσουμε λοιπόν τώρα με την Κομισιόν και φυσικά θέλουμε να μάθουμε πώς πηγαίνουν οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς ε, και πώς είναι ε, η κατάσταση, πώς έχει η κατάσταση. Τι να περιμένουμε, ότι θα λήξει η συγκεκριμένη εξαίρεση ή τι θα γίνει μετά την 1η Μαΐου. Ε, ένας από τους ε, ειδικού ε, της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει πάνω σε αυτό. Και αυτό φυσικά σχετίζεται με αρκετά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα την νομιμότητα αυτής της πράξης 232 ε, και της, ε, και της 231 που επίσης επικαλείται ο ε, πρόεδρος. Πιστεύω ότι, έχω, ότι δεν λαθάνω, είναι η 231 του 61 Πρόκειται για μια παλαιά εμπορική πράξη και δεν συνάδει ε, με τους κανόνες του ε, ΠΟΕ. Ε, ποια είναι η θέση της Κομισιόν πάνω σε αυτό. Δεύτερον, η Κομισιόν ανακοίνωσε μία προσφυγή κατά αυτών των μέτρων της, των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΠΟΕ και ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε και γι' αυτό. Τρίτον, τι αντιμέτρα θα υπάρξουν σε περίπτωση που από την 1η Μαΐου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το, ε, αυτούς τους δασμούς 25% ε, στον χάλιβα και 10% στο αλουμίνιο και αν θα ε, υπάρχει ε, πιο έντονη ε, σχέση με άλλους τέρους όσον αφορά τα συγκεκριμένα αγαθά. δεν θα αναφερθώ στο TTIP διότι δεν νομίζω ότι ταιριάζει αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με ξανακαλέσετε στην Επιτροπή σας για να σας κάνω μια ενημέρωση για τα αμερικανικά μέτρα για το χάλιβα και το αλουμίνιο. Μετά από το τελευταίο θέμα που συζητήσαμε για τις σχέσεις με την Κίνα, έχει ενδιαφέρον ότι αν το δούμε και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι υπάρχει, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση να γίνεται μετά από τη συζήτηση που κάναμε για την Κίνα και τα πράγματα έχουν ως εξή. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα πριν από το Μάιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποκλείσει προσωρινά έξι εμπορικούς εταίρους από τα μέτρα για το Χάλιβα, τον Καναδά, το Μεξικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Νότιο Κορέα. Και μέχρι σήμερα έχουν μια συμφωνία με την Νότια Κορέα και με, για τους άλλους πέντε συνεχίζονται οι συζητήσεις. Τι προβλέπουμε εμείς ότι η διοίκηση Τραμπ στα τέλη της εβδομάδας θα εξετάσει όλες αυτές τις περιπτώσεις αυτών των εταίρων και τις επαφές με αυτούς ώστε να αποφασίσει αν θα παρατείνει ε, την, ε, το μέτρο αυτό ή αν θα δώσει μόνιμη εξαίρεση ή αν δεν θα εξαιρέσει πλέον αυτές τις χώρες από τους δασμούς για τις ε, εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου που τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν στον κόσμο που εξάγουν προς τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή ε, υφίστανται αυτούς τους δασμούς. Εμείς ε, στις επικοινωνίες μας με τους Αμερικανούς φίλους και εταίρους έχουμε κοινοποιήσει πέντε άξονες που χαρακτηρίζουν την απάντησή μα. Εμεί δεν συμβάλλουμε στην πλεόνασμα παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί την τελευταία πενταετία. Δεν είμαστε εμεί ε, πηγή μεταφόρτωσης ε, χάλιβα που παράγεται με αθέμητο τρόπο σε τρίτες χώρε και που διέρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να καταλήξει στι Αμερικανικέ αγορέ. Έχουμε πολύ ισχυρή νομοθεσία προστασίας από τις μεταφορτώσεις δρούμε εμείς οι ίδιοι κατά των αθέμητων εισαγωγών χάλιβα και από την Κίνα. Δεν ρίχνουμε φθηνό χάλιβα στην Αμερικανική αγορά. Οι μέσες μας τιμές ε, χάλιβα που, εξ, ε, που εξάγεται στις ΗΠΑ είναι αρκετά ψηλές, διότι εξάγουμε χάλιβα και αλουμίνιο υψηλής ποιότητας που χρειάζεται η Αμερικανική οικονομία. Συμμετέχουμε ενεργά στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Χάλιβα που έχει ως στόχο την ε, εκπόνηση νέων κανόνων, καλύτερων κανόνων, καλύτερο έλεγχο των επιδοτήσεων και μείωση της παραγωγής ε, μέσω της συνεργασίας όλων των χαλιβοπραγωγών ε, σε όλο τον κόσμο και μετά εδώ και δεκαετίες είμαστε αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο τη επικοινωνία μα λοιπόν με τι ΗΠΑ έχουμε πει ανεπιφύλακτα ότι θεωρούμε ότι αιτιολογείται απόλυτα η εξαίρεση που πρέπει να χορηγηθεί μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους ε, δασμούς αυτούς. Επίσης τους έχουμε ενημερώσει ότι πιστεύουμε πως δεν αιτιολογείται έρευνα σε θέματα εθνικής ασφάλειας, λόγω θέματων εθνικής ασφάλειας. Ο Επίτροπος μας ε, ε, μίλησε σε διάφορους συναδέλφους ε, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο λέγοντας ότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ε, λόγος αιτιολόγησης τέτοιων περιορισμών εξαγωγής για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εμείς θεωρούμε, όπως εξήγησαμε, ότι αυτά τα μέτρα υιοθετούνται κρυφά και βάσει αυτής της νομικής βάσης ζητάμε ή ΙΠΑ να ανταποκριθούν ε, για την προστασία των δικαιωμάτων μας στο σύστημα του ΠΟΕ. Υπάρχουν τακτικές λοιπόν επαφές μεταξύ ημών και των Πολιτειών, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο επιτρόπου δηλαδή. Εμεί έχουμε διαβιβάσει διάφορα ηχηρά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι αμφισβητούμε την ομιμότητα των μέτρων αυτών που έλαβαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το δεύτερο είναι ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε για την εξέβρεση λύσεων που δεν επιτρέπονται δυνάμει των κανόνων του ΠΟΕ. Ε, διάφορες εθελοντικού περιορισμούς εξαγωγών και διάφορες τέτοιε διευθετήσει ε, που ήταν συνήθες το 1980 και το 1990 αλλά που πλέον δεν επιτρέπονται δυναμικά ε, συγκεκριμένων συμφωνιών του ΠΟΕ όπως λειτουργεί σήμερα. Η γραμμή που ακολουθούμε εμείς λοιπόν στην επικοινωνία μας με τις ΗΠΑ είναι ότι ζητάμε απόλυτο εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτούς τους δασμούς όσον αφορά το χάλιβα και το αλουμίνιο. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε εν ώψη της 1ης Μαΐου βάσει των πέντε επιχειρημάτων που μόλις σας παρουσίασα. Διότι η Ευρώπη ουσιαστικά λέμε εμεί ότι δεν είναι κομμάτι του προβλήματος αλλά κομμάτι της λύσης αυτού του προβλήματος της, ε, του πλεονάσεως παραγωγής. Από την αρχή μάλιστα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Από όσο γνωρίζουμε, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από τον ε, Πρόεδρο προσωπικά. Οπότε την 1η Μαΐου θα δούμε τι θα κάνουμε, ποια θα είναι η αντίδρασή μας ε, ανάλογα με το ποια από τις τρεις επιλογές θα κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρόεδρος. Δηλαδή αν θα είναι η επιλογή μόνιμη εξαίρεση, προσωρινή παράταση της υπάρχουσας εξαίρεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιβολή των δασμών στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από αυτές τις τρεις ε, δυνατότητες, εμείς ε, εξακολουθούμε να επιδιώκουμε την προστασία των δικαιωμάτων μα Αυτό πρέπει να το επιδιώκει κανείς ενεργά στο σύστημα του ΠΟΕ. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Έχουμε λοιπόν ε, καταρτήσει μια λίστα προϊόντων. Αυτό που ονομάζουμε λίστα επανεξισορρόπησης δεν είναι αντίμετρα, αντίπεινα. Βασί διαδικασιών του ΠΟΕ, αν αποσύρει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβαση στην αγορά ένας εταίρος, έχει κάνει το δικαίωμα να αποσύρει αντίστοιχο όγκο, ώστε να επέλθει μια νέα ισορροπία στη σχέση μεταξύ των δύο μερών. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτές τις λίστες ως λίστες επανεξισορρόπησης. Λίστες που αποσκοπούν στο να προστατεύσουν εμάς ε, Έχουμε συμφωνήσει ομόφωνα ήδη από την περασμένη Τρίτη με τα κράτη-μέλη για τη λίστα αυτή. Εγκρίθηκε δηλαδή και τώρα ε, περνάει από τις εσωτερικέ μας διαδικασίες για να εγκριθεί εδώ και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί στον ΠΟΕ μέχρι τις 22 Μαΐου. Αν δεν κάνω λάθο πρέπει να έχει γίνει μέσα σε 60 ημέρε, ώστε να, να διαφυλαχθούν τα δικαιώματά μα. Ρωτήσατε επίση, κύριε Πρόεδρε τι κάνουμε για να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή αγορά από το πλεόνασμα χάλιβα που θα εμφανιστεί στην παγκόσμια αγορά απλά διότι δεν θα μπορέσει να μπει στην αμερικανική αγορά από τις 23 Μαρτίου έχει συμβεί αυτό. Έχουμε ξεκινήσει έρευνες ε, διασφάλισης της παρεκτροπής ε, του εμπορίου κάτι που αφορά διάφορα προϊόντα ουσιαστικά και που όλα τα προϊόντα για τα οποία έχει επιβληθεί περιορισμό εισαγωγών στι ΗΠΑ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο αυτέ οι εξαιρέσει, ε, αυτέ οι αποκλεισμοί, συγγνώμη, ε, θα συνεχιστούν. Αν δεν συνεχιστούν, εκεί φυσικά ε, θα υπάρξει όλο και περισσότερο χάλιβα, ο οποίο θα εμφανίζεται στι ευρωπαϊκέ αγορέ, θα περεκτρέπεται προ τι ευρωπαϊκέ αγορέ και εμείς ε, κοιτάμε τα νούμερα σε μηνιαία βάση, διότι τα μέτρα διασφάλισης μπορούν να εφαρμοστούν μόνο εφόσον υπάρξει αύξηση των εισαγωγών. Το παρακολουθούμε λοιπόν στενά. Αποτελέσματα βλέπει κανείς διαφορετικά ανάλογα με τη χρονική στιγμή. Στην αρχή ε, παρακολουθούσαμε την εκτροπή ε, συγκεκριμένου αριθμού, περιορισμένου αριθμού εμπορευμάτων και μετά παρακολουθούμε τα εμπορικά νούμερα με στους επόμενους μήνες για να δούμε κατά πόσο απαιτείται περαιτέρω μέτρα προστασίας ε, για άλλα προϊόντα. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Απλά οι εργασίες αυτές βρίσκονται υπό εξέλιξη. Θα έχουμε συναντήσεις και αυτή τη βδομάδα με τα τη μελη μας, αν δεν κάνω λάθος, και θα κάνουμε κάποιες αρχικές προσωρινές ε, αξιολογήσεις ε, αρχές Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Ε, το άλλο που ρωτήσατε κύριε Πρόεδρε ήταν τι γίνεται με τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Εμείς αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις που ζήτησε η Κίνα να γίνουν με τη ΣΥΠΑ με την επιφύλαξη οποιονδήποτε αποφάσεων εμεί θα λάβουμε αργότερα το κατά πόσο θα συμμετέχουμε ως τρίτο μέρος ε, στη ε, διαφορά αυτή ή αν θα ξεκινήσουμε δική μας ξεχωριστή διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω διάφορες, ε, διάφορα αιτήματα, τέσσερα, πέντε άνθρωποι ζήτησαν το λόγο και έχουμε μόνο πέντε λεπτά. Ένα λεπτό, λίγο λιγότερα από ένα λεπτό καθένας. Ένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Η Επιτροπή θέλει να συζητήσει τα προβλήματα με τις ΕΙΠΑ. Ποια θέματα θα ε, χρησιμοποιήσετε ως ε, επιχείρημα ε, για να υπερασπίσετε το εμπόριο αυτό. Και μετά, ο Μακρόν βρίσκεται στη ΣΥΠΑ αυτή τη βδομάδα. Θα θέσει το ζήτημα, είμαι σίγουρη θα υπάρξουν κάποιε επαφέ μεταξύ του Μακρόν και τη Κομισιόν όσον αφορά αυτέ Τι εξελίξει. Ε, Τιτσιάνα Μπεγκίν. Ευχαριστώ πολύ Τιτσιάνα Μπεγκίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακόμα περισσότερο από του δασμούς αυτό που βλάπτει είναι η αβεβαιότητα. Γιατί έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν προγνωστικά για το μέλλον. Εγώ νομίζω ότι πάντως ότι παίζουμε το δικό τους παιχνίδι με τις με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Ε, αυτή είναι από θέσεως ισχύω, εμείς είμαστε διαιρημένοι. Ε, έχουν αυτή το περίστροφο πάνω στο τραπέζι. Και εμείς έχουμε μάλλον διστακτική αντίδραση όσον αφορά τους δεσμούς. Βεβαίω, και δεν ωφέλει κανένα εμπορικό πόλεμος. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος να πάμε με τα νερά του. Δεν είναι ο μόνος δρόμος η διπλωματική λύση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε αναμέτρηση δυνάμεων. Πιο δυναμικά δηλαδή. Επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πολιτικό διαβάσαμε για τις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ. Για το ότι πώς προχωράει η υπόθεση τι, σιγά σιγά, τι γίνεται κατά της πολιτικής Τραμπ, τι είπε η κυρία Μάλμστρομ, που δεν θέλει να ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. για να τα λέμε όλα, υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν πάρα πολλέ αντιρρήσεις από πλευράς ε, διατροφικής ασφάλεια και ε, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Δεν ε, υπάρχει κάποιο ε, πίεση όσον αφορά τα πρότυπα. Δεν ξέρω πώ θα πάνε οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομη ερώτηση όπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα γίνει να πάμε στο κακό σενάριο. Και τελικά, εάν επιβιωθούν αυτοί οι δασμοί. Και αν τελικά χτυπηθούν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε λόγω των νέων αυτών δασμών. Μπορούμε να αξιώσουμε αποζημίωση για αυτές τις εταιρείες που θα πληγούν από τους δασμούς. Και εγώ, κ. Σόλτς, να υποβάλω μια ερώτηση Πέραν αυτών των οποίων είπαμε την στο Στρασβούργο όσον αφορά το πολυμερές φόρουμ του Χάλιβα, με τι χρονοδιάγραμμα, τι μέτρα προγραμματίζεται. Γιατί είπε και ένας ότι πάμε για Ιούλιο, Αύγουστο και ίσω πιο νωρίς και για Μάιο. Οπότε τι λογαριάζει να κάνει η Κομισιόν. Εγώ να σας πω τα εξής, να σας τα πω στα Ολλανδικά. Καταλάβαμε πριν την εβδομάδα ότι ήρθε η ώρα να έρθουμε σε επαφή και να τα συζητήσουμε με του Αμερικανούς και όχι μόνο με αυτού, όσον αφορά το ότι πρέπει να υπάρξει μια ανοιχτή εμπορική πολιτική. Α τελικά όμω. δεν έχει δημορφωθεί κάποια ε, κατάλληλη ψηφία αυτό που θα κάνουμε από πλευρά Επιτροπή ή Κοινοβουλίου. Πώ το καταλάβατε ποτέ, πώ τα Ναι, ναι, και εγώ θα σα ρωτήσω, ε, ε, ε, τι, τι πιθανότητες έχουμε για εξελίξει στην 1η Μαΐου. 60, 40, 50. 50 να σα πω πρώτα, λέει η Κομισιόν. Δεν μπορώ να ρισκάρω. Ο υπάλληλο είμαι. Δεν θα τολμήσω προγνωστικά. Για αυτά όλα που μας ρωτήσατε, εμείς σας λέμε ξεκάθαρα. Εμείς θέλουμε χωρίς καμία προϋπόθεση και περιορισμό να εξαιρείται από αυτούς τους δασμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη διαπραγματεύσεις. Ε, που εξελίξει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται εδώ σε κοινοβούλια και σε συμβούλια. Αλλά τέλος πάντων αυτό θα ακολουθήσουν. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να αποσπάσουμε αυτή την ε, εξαίρεση σαν καθαρή λύση. Και νομίζω αυτό καλύπτει πολλούς από εσά που υποβάλλατε ερωτήσει. Επίσης, Όχι, όχι. Δεν θέλουμε να πάμε για αναθεώρηση του TTIP. Ούτε εμείς, ούτε και οι Αμερικανοί. Τώρα γι' αυτό που ρώτησε ο κύριος Βίγκλη, δεν θα γίνει να τελικά το κακό σενάριο. Ε, σε αυτή την περίπτωση, ε βέβαια και θα προσπίσουμε τα δικαιώματά μας. Και θα συνοηθούμε με το Συμβούλιο και με εσάς για το πώς θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτά τα οποία προβλέπονται από τον ΠΟΕ. Αν χρειαστεί, δικαιούμεθα να λάβουμε μέτρα. Όμως θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να σκεφτούμε το τι θα κάνουμε. Αλλά βέβαια θα υπάρχουν και αρνητικέ συνέπειε. Γιατί αν δεν υπάρχουν κάποιε επαναστατικέ αλλαγέ, πρέπει να ζούμε τη σύμβαση άλλα μέτωπα Φερρυπίν όσον αφορά τη θωράκιση των διεθνών κανόνων για το πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποιες κρατικές ε, εταιρείε που δρούν στο, στη διεθνή εμπορική σκηνή και έχουμε τώρα το 301 του ΠΟΕ. Γιατί σας τονίζω ότι βλέπονται πολλά διαφορετικά πράγματα σε αυτή την ε, πρόστριβη και πάρα πολλά παίζονται για τη ΣΥΠΑ. Τώρα για το 6. Και τελειώσαμε πριν πάμε στο 7 να καλωσορίσουμε τον Αλεξάνδρ Γκάμπελιτ, το νέο μέλος της Επιτροπής μας. Καλή επιτυχία, καλή δουλειά εδώ στην Επιτροπή μας. Πάμε τώρα στο σημείο παραδείγματων 7. Το κοινό έργο, ΙΜΚΟ και ΙΤΑ, τα σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Έχουμε μαζί μας την ε, πρόεδρο της ε, ΙΜΚΟ, γίνεται ε, με βάση τον κανονισμό 55. Ε, κάθε συνάντηση θα έχει διαφορετική ε, ημερήσια διάνταξη και θα έχουμε μία τελική έκθεση